Ε, και... Συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Το επόμενο, το επόμενο σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση με θέμα ευθυγράμμιση προς τη συνθήκη της Λισαβόνας πρώτος εισηγητής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης Πέθρου του Παϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πάολο Ντεκάστρο. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η συνθήκη τη Λισαβόνα καταργεί το παλιό σύστημα τη επιτροπολογία και το αντικαθιστά με μια δομή δύο επιπέδων που βασίζεται στι ε, πράξει κατευθυνότηση, και σε εκτελεστικές πράξεις που αποκλείουν παντελώς το Κοινοβούλιο σε κάθε φάση της έγκρισής τους. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να ευθυγραφίσουμε το, το ζήτημα με τις νέες απαιτήσει. Υπάρχουν τρεις βασικοί κανονισμοί, τους οποίους πρόεδρε θα θίξω ομού σε τις άμεσες πληρωμές, την ανάπτυξη της υπέτρου και την κοινή οργάνωση αγορών. Οι προτάσεις ε, της ε, Κομισιόν μας φάνηκαν ε, εξορροπημένες και οι αλλαγές που έκανε η Επιτροπή Γεωργίας ήταν πραγματικά ελάχιστες. Ειδικά σε ό,τι φορά τις άμεσες πληρωμές και τις, για τις πράξεις του κατεξοδότηση θα πρέπει να χορηγούνται μόνο σε ορισμένε περιπτώσει, όπου ενδέχεται να υπάρχουν και αρνητικέ επιπτώσει για του Γιώργου. Επίση, θεωρήσαμε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη για την κοινή οπτική πολιτική σε ζητήματα προπολογισμού, η δημοσιονομική πειθαρχία θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλέον δίχω τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου. Να διατηρήσει, λοιπόν το άρθρο 11 ε, αμετάβλητο που προβλέπει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει μετά ο πρόεδρος της Κομισιόν. Αυτό θα αποτελούσε παραβίαση των ε, αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, η Κομισιόν θεωρούμε ότι έκανε μια σωστή κατανομή ανάμεσα στις γενικότερες διατάξεις που περιέχουν συμπληρωματικά στοιχεία και αφορούν τις κατευθυντικές του πράξη και πιο τεχνικά ζητήματα που αφορούν στην διακριτική, διακριτική μεταχείριση που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και εδώ πρόκειται για εκτελεστικές ε, πράξεις. Τώρα για την κοινή οργάνωση αγορών βλέπουμε ότι υπήρξε μεγαλύτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στο άρθρο 43 3 τις συνθήκες ε, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συνθήκη αυτή προβλέπει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Κομισιόν να υιοθετήσει τα σχετικά μέτρα για τον καθορισμό των τιμών και για τους ποσοτικούς περιορισμούς. Πρόκειται για μια ε, ε, εξαίρεση σχέση με παραφοβείο του αυτού άρθρου για την προσφυγή στην ε, ε διαδικασία, νομοθετική διαδικασία. Τώρα, προκειμένου για εξαίρεση, το άρθρο 43.3 θα πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο περιοριστικό. Δηλαδή μόνο όταν υπάρχουν διατάξεις που δεν αφορούν πολιτικές θεμελιώδεις αποφάσεις που θα πρέπει να ε, εφαρμοστούν σύμφωνα με το 43.2. Θεωρούμε πως η πρόταση της Κομισιόν δεν ερμηνεύει με τρόπο επαρκώς περιοριστικό το άρθρο 43.3. Ο ορισμός των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για τον καθορισμό των ενισχύσεων, για τις επιστροφές, τις εξαγωγές, για τις ελάχιστες τιμές των εξαγωγών θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του νομοθετικού σώματος του Κοινοβουλίου δηλαδή και του Συμβουλίου ενώ η Κομισιόν θα, θα ασχολείται με τον καθορισμό των τιμών μέσω κατεξοδότηση πράξεων. Όταν, εγκριθούν, λοιπόν, αυτά, όταν εγκρίθηκαν αυτά τα στοιχεία στην Επιτροπή Γεωργία, αρχίζαμε να διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν να κανορθώσουμε να πετύχουμε, Πρόεδρε, μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ε, το κατεπήγον ε, οφείλεται στην επικείμενη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική που θα θελήσαμε να μην επηρεαστεί από περίπλοκε διαπραγματεύσει πάνω σε θέματα θεσμική φύση αλλά παρά την διαθέσιμότητά μας για διαπραγμάτευση και να ε, παραχωρήσουμε κάτι σε σχέση με την αρχική μας θέση και παρά την δραστήρια στάση της ε, Πολωνικής και της Δανικής Προεδρίας δεν καταλήξουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό. Άρα η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να ενεργεί άμεσα και να ε, τηρηθούν οι νέες εξουσίες του Κοινοβουλίου. Βασικά εμπόδια τα βρήκαμε ε, με το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο που ήθελε να καταργήσει τις ε, κατοξιότητες πράξεις, ακόμα και όταν αυτές είναι νομοθετικά υποχρεωτικές για να τις εφαρμόζει με εφαρμοστικές πράξεις προκειμένου να αποκλειστεί το, Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας, διότι σημαίνει να παρελθούν τις νέες ε, εξουσίες που μας χορηγεί η συνθήκη. Το ένα άλλο στοιχείο που κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη διαπραγμάτευση ήταν η στάση της Κομισιόν που ε, από μια θέση που προσέγγιζε αυτή του Κοινοβουλίου μετακινήθηκε στις, ε, προς τις του Συμβουλίου και μας άφησε μόνους για να υποστηρίξουμε τις ε, τα άρθρα τη συνθήκη. Τώρα έχουμε μπροστά μα την μεταρρύθμιση ΚΑΠ. Ζητήσαμε από την Ολομέλεια, μάλλον θέλουμε να ζητήσουμε την Ολομέλεια να επιβεβαιωθεί η ψηφοφορία στην Επιτροπή Γεωργία για να έχουμε μεγαλύτερη ισχύ όταν θα διαπραγματευτούμε τη μελλοντική ε, αγροτική πολιτική. Μόνο υποστηρίζοντα τι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου, θα μπορέσουμε να τηρήσουμε και να σεβαστούμε στην Λισαβόνα και να καταστήσουμε την ΚΑΠ του μέλλοντο πιο δημοκρατική και πιο κοντά στου πολίτε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Επόμενος εισηγητής είναι ο συνάδελφος κύριος Τζιωβάνι Λαβία και έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Μετά από τη θέση ισχύ της δίκης Λισαβόνας, ε, η ε, δράση ευθυγράμμισης ε, στις νέες συνθήκες της στις ανάγκες της συνθήκης αφορά στο θέμα των ε, διατάξεων που εθέτησε το, ε, η Κομισιόν. Αφού, εξετάσαμε την πρόταση της Κομισιόν για τις δύο κατηγορίες των πράξεων, ε, τα άρθρα 290 και 291, εντοπίσαμε ζητήματα για τα οποία προβλέπονται κάποιες προϋποθέσεις. Εξετάσαμε την πρόταση σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις για τις εκτελεστικές πράξεις. Στην Επιτροπή Γεωργίας προτείναμε και εγκρίναμε κάποιες προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την ανάθεση εξουσιών, την παράταση των προθεσμιών, τις διαδικασίες της Επιτροπής και τις πρακτικές μετά από έγκριση του, του Προεδρείου το Μάρτιο 2011 και τον κανονισμό το σχετικό για τον έλεγχο από πλευράς κρατών των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών που ανατίθεται στην Κομισιόν. Μεταξύ των διαφωνιών που είχαμε ανάμεσα με το Συμβούλιο αναφέρομαι στις εκτελεστικές πράξεις ε, όπου σύμφωνα με τις συνθήκες αυτό θα ήταν το πιο ε, εύλογο μέσον και πλέον κατάλληλα αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραιτηθεί από το να ασκεί έλεγχο σε ζητήματα τόσο ευαίσθητα και σημαντικά όπως τη διαφάνεια, άρθρο 40α ή τις κυρώσεις των δικαιούχων. Αυτό λοιπόν το ζήτημα των ευθυγραμμίσεων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και αφορά στην συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Σύμφωνα με τις διαθρωμένες αρμοδιότητες που θα έπρεπε να συγκλίνουν προς την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Οι πλειοψηφίε που απαιτούνται στο Συμβούλιο για να ε, περιοριστεί η εφαρμογή των ε, εφαρμοστικών πράξεων είναι περιορισμένη και άρα δεν είναι αιτιολογημένη. Αν διατηρηθεί θα, θα είναι ένα περιττό εμπόδιο στη μεταρρύθμιση κοινής αγροτική πολιτικής. Να πω επίσης πως προτείναμε κάποια στοιχεία προκειμένου να βελτιωθεί, αλλά δεν έτυχαν τις έγκρισης της Κομισιόν και του Συμβουλίου και ως εκ τούτου θα αποτελέσουν τμήμα διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της οριζόντιας μεταρρύθμισης του ΚΑΠ. Η έλλειψη συμφωνίας ε, σε ό,τι αφορά την ευθυγράμμιση του οριζόντιου κανονισμού μας ανάγκασε να ζητήσουμε αυτήν την ψήφο από την Ολομέλεια για να αποκτήσουμε όπως είπε ο πρόεδρος Κάστρο μια μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ ε, πάνω στο ζήτημα αυτό απέναντι στο Συμβούλιο. Τώρα, τόσο αυτό το ζήτημα όσο και τα άλλα τα οποία εξετάσαμε μέχρι τώρα ήταν πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο που για πρώτη φορά μέσω της συναπόφασης εμπλέκεται σε ό,τι φορά στον προσδιορισμό και διατύπωση της νέας γεωργικής πολιτικής. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα απλό, απλά μεταφοράς όπως πολλοί είπαν, αλλά για μια συνειδητοποίηση από τους αδέρφους στην Επιτροπή Γεωργίας σχετικά με τη λειτουργία της ΚΑΠ μέχρι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να προχωρήσουμε. Για να πω κάτι ακόμα, μέσω μιας μακράς πορείας ε, των τριμερών διαλόγων προσπαθήσαμε να πετύχουμε μια ε, συμφωνία σε αυτή την ευθυράμιση προς τη συνδίκη Λισαβόνας. Χάσαμε χρόνο. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στο μέλλον. Yeah. Σειρά εισηγητή είναι ο συνάδελφο κύριο Μάρτιν Χόισλινγκ, τον οποίο τον καλώ στο βήμα επίση για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, όπω είπαν και οι προηγούμενοι και για την βιολογική γεωργία, πρέπει να προχωρήσουμε σε πρώτη ανάγνωση αυτό είναι κρίμα, αλλά κάναμε τρεις τριμερείς διαλόγους όπου δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος. Ήταν βέβαια φιλική ατμόσφαιρα, αλλά στα κέρια θέματα δεν επετέφθη συμφωνία. 1η Ιουνίου πέρσι στην Επιτροπή Γεωργίας έγινε δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία η έκθεση για την προσαρμογή. Μετά άρχισαν οι διαπραγματεύσεις υπό Πολωνική Προεδρία και μετά υπό Δανέζικη Προεδρία και συνεχίσαμε βέβαια τις διαπραγματεύσεις. Δεν προχωρήσαμε σε δύο θέματα. Πρώτον στα προϊόντα και ουσίες και για τους σχετικούς ισχυρισμούς, claims, δεν μπορέσαμε δηλαδή εκεί να πετύχουμε συμφωνία και δεν βασιστήκαμε μονάχα στις δικές μας απόψεις ζητήσαμε να ψηφίσει και η Νομική Επιτροπή γνωμοδότηση και μας είπε καθαρά ότι πρόκειται για νομικές πράξεις που πρέπει να είναι κάτω Πρόκειται για το άρθρο 290. Εκεί ρυθμίζεται η υπόθεση αυτή και είναι σαφές ότι πρέπει να πρόκειται για κατεξουσιοδότηση πράξης. Όχι τι ρύθμιση είναι, αλλά ότι η ρύθμιση αυτή είναι δεσμευτική και ότι είναι ομοιόμορφα δεσμευτική για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν ό Κοινοβούλιο κατανοούμε τη θέση του Συμβουλίου ότι επιθυμεί να εμπλέκεται και το τονίσαμε κατά επανάληψη στις διαπραγματεύσεις ότι έχουμε κατανόηση κάναμε άλλωστε και συμβαστικές προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή είπαμε δηλαδή να περιληφθούν οι πραγματογνώμονες από τις εθνικές ε, αντιπροσωπείες να βάλουμε και τις ουσίες στα λεγόμενα basic acts και είπαμε ότι αυτά μπορούν να γίνουν δεκτά. Είναι κατανοητό δηλαδή διότι υπήρξαν δύο αλλαγές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Είναι επομένω λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Τώρα, για όλη αυτή τη διαδικασία θα συμφωνήσω με τον ε, κύριο Δεκάστρο ότι η Κομισιόν άλλαξε την στάση της διαρκούντος του τριμερούς διαλόγου για τις ε, κατεξουσιώδεις πράξεις. Εμείς δεν το κατανοήσαμε αυτό. Μετά μας έγινε μια αόριστη πρόταση ότι θα ενημερωνόμαστε όταν θα επίκυνται αλλαγές. Αυτό βεβαίως για μας δεν είναι αρκετό. Εμείς έχουμε το δικαίωμα να επιμείνουμε σε κατεξουσιοδότηση πράξης και αυτή τη θέση μας θα ενισχύσουμε και στην πρώτη ανάγνωση και ελπίζουμε η Κομισιόν να έλθει να υποβάλει πλέον πρακτικά εφαρμόσιμες προτάσεις που να μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε τη διαπραγματεύσεις υπό Κυπριακή πλέον Προεδρία. Ο κύκλος των εισηγητών ολοκληρώνεται με την ε, ομιλία του συναδέλφου κ. Καπούλα Σάντος, ομοίως για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεσή μου αφορά στους ελέγχους εκ μέρους των κρατών μελών ε, σχετικά με πράξεις ε, που αποτελούν μέρος του συστήματος χρονοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγύησεων. Πρόκειται για την ευθυγράμμιση στον κανονισμό για τις ε, κατεξόρυση πράξεις, για τις εκτελεστικές πράξεις έχουν προβλεφθεί κάποιες ε, διατάξεις με βάση τον κανονισμό για τον ε, άσκηση ελέγχου από πλευράς Κομισιόν. Για τις της πράξεις ε, βασιστήκαμε στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα όργανα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να βεβαίωσει αυτή την στάση στην αυριανή ψηφοφορία. Αυτή η ψηφοφορία θα πρέπει, μάλλον η υπεψήφιση θα πρέπει να είναι ευρύτερη δυνατή ή δυνατόν ομοφωνία. Θα ήθελα να κάνω έκκληση προς το Κομισιόν και το Συμβούλιο για μια ε, αυστηρή εφαρμογή της Θήκης Λισαβόνας για να πετύχουμε την πρόοδο που επιθυμούμε στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης ΚΑΠ. Ο χρόνος πιέζει. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μετατρέπει την παλαιά επιτροπολογία και προβλέπει μια σαφή διάκριση ανάμεσα σε, σε εκτελεστικές πράξεις και την δυνατότητα ε, ανάθεσης ε, ενός ενισχυμένου δικαιώματος ε, άσκησης βέτο και ανάκλησης της ανάθεσης από πλευράς του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν συνεχίζει να διατηρεί τις εξειδικευμένες επιτροπές και προβλέπεται διαβούλευση με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για την επεξεργασία των ε, κατοξιδότηση πράξεων. Χρειάζεται να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις κατοξιδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις έτσι ώστε τα όρια ανάμεσα στα, στις δύο αυτές πράξεις να αφήνουν περιθώρια ερμηνείας. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο αποκτά νέες αρμοδιότητες. Δεν ζητώ το Κοινοβούλιο να υποκαταστήσει το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κομισιόν, αλλά διεκδικούμε για το Ευρωκοινοβούλιο ένα δικαίωμα ελέγχου στο πλαίσιο της νέας επιτροπολογίας. Όλα λοιπόν θα πρέπει να είναι ανάλογα και αναλογικά συγγνώμη με το... Κύριε Τσόλος, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία και πάλι να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή Γεωργίας και το σύνολο των εισηγητών για τη σημαντικότατη εργασία που έγινε. Αυτές οι προσπάθειες μας βοηθήσανε να προχωρήσουμε με το φάκελο της ευθυγράμμισης και θέλουμε όλοι να καταλήξουμε. Όπως ξέρετε, όλη αυτή η άσκηση της ευθυγράμμισης είναι πρώτα πολυτεχνικό θέμα, όπως άλλωστε αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε και από τα σχόλια των εισηγητών. Είναι περίπλοκο νομικά, αλλά είναι και μία άσκηση πολύ ευαίσθητη πολιτικά ειδικότερα για το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και για όλα τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή της ΚΑΠ. Έχω απόλυτη συνείδηση της πολιτικής σημασίας λοιπόν της συζήτηση για την ευθυγράμμιση στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Δεκάστρο, οι συζητήσεις ξεκινήσαν κάτω από Ουγγρική Προεδρία και συνέχισαν ε, εδώ και ένα χρόνο. Κάποια στιγμή κοντέψαμε να συμφωνήσουμε, αλλά τελικά βρεθήκαμε σε αδιέξοδο μετά τον τελευταίο τρίλογο κάτω από την Πολωνική Προεδρία. Στη συνέχεια η Ιδανική Προεδρία αποφάσισε να βάλει το τμήμα της ευθυγράμμισης στη συζήτηση για την ΚΑΠ και να έχουμε και ξεχωριστή συζήτηση για την ευθυγράμμιση. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι σαφής. Ε, το έχω πει πολλές φορές στην Επιτροπή Γεωργίας, αλλά το επαναλαμβάνω και εδώ. Πάντα θέλησα να προασπίσω τα προνόμια του Ευρωκοινοβουλίου όπως προκύπτουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας για όλο το πακέτο της ευθυγράμμισης για να έχουμε μια ισορροπημένη κατανομή Οπότε υπήρχε μια γκρίζα ζώνη και κάθε φορά που ήταν εφικτό νομικά, το υπογραμμίζω αυτό, προτιμούσα μια προσέγγιση που έδινε δυνατότητα και στους δύο θεσμούς να παίξουν το ρόλο τους. Ε, προτιμούσα την αυστηρή εφαρμογή του 43-3 της συνθήκης της Λισαβόνας, δίνοντας ε, το προβάδισμα στις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Γι' αυτό και για τις άμεσες ενισχύσεις έδωσε ε, ρόλο αν θέλετε στην δημοσιονομική πειθαρχία και στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο και στον προσδιορισμό των μονίμων βοσκοτόπων επίσης προτίμησα τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πολλά παραδείγματα μπορώ να σας δώσω ακόμη και στον τομέα των κυρώσεων. Σας παρακαλώ να τα δείτε λεπτομερώς για να δείτε, για να διαπιστώσετε ότι η Κομισιόν πραγματικά κατέβαλε προσπάθειες για να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Αλλά από αυτό το σημείο εκκίνησης που δίνει ένα ενισχυμένο ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο δεν συμφώνησε πάντα και βεβαίως χρειάστηκε να βρούμε και συμβιβασμούς. Γενικά όμως από αυτό το σημείο εκκίνησης που σας προσδιορίσα, το γενικό πακέτο των συμβιβασμών σε κάθε άσκηση ευθυγράμμισης ενίσχυσε τα προνόμια του Ευρωκοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε αυτή η άσκηση ευθυγράμμισης να αδικήσει τις επί ουσίας συζητήσεις για την κάπου είναι σημαντικές για όλους μας. Θεωρώ αυτή την ψηφοφορία σαν σήμα προς αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Τώρα, ειδικότερα όσον αφορά την οργανική γεωργία, τα βιολογικά προϊόντα. Ε, δεν έχουμε ακόμη συμφωνήσει για τα πιο ευαίσθητα σημεία, δηλαδή τη διαδικασία αδειοδότησης των ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βιολογική γεωργία. Αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείται ότι η αδειοδότηση μη ορισμένων ουσιών ή τάξεων ουσιών έχει πολιτικό χαρακτήρα μέσα στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Συνεπώς, δεν θέλετε να αποκλειστείτε από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί αυτών των ουσιών. Υποστηρίζω την προσέγγισή σας, τη θέση σας. Νομίζω όμως ότι οι δισταγμοί σας συνδέονται με την σημερινή διατύπωση του κανονισμού για τη βιολογική καλλιέργεια Πράγματι τα κριτήρια εκεί μπορούν να βελτιωθούν, να προσαρμοστούν. Μπορώ ακόμη να αντιληφθώ ότι πολλοί από εσά πιστεύετε ότι είναι ευκταίο να επικαιροποιηθούν και να εξειδικευθούν αυτά τα θέματα κάθε φορά που είναι εφικτό. Ακριβώς αυτό προτιθέμεται να κάνουμε η Κομισιόν ενέκρινε μια έκθεση βάσει της κεκτημένης εμπειρίας για την εφαρμογή των κανονισμών βιολογικής καλλιέργειας από το 2009. Αυτή η έκθεση αποτελεί την πρώτη φάση μιας συζήτησης γύρω από το θέμα της βελτίωσης του νομικού πλησίου για τη βιολογική παραγωγή. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία αξιολόγηση, μία μελέτη επιπτώσεων και το θέμα της επικαιροποίηση των κριτηρίων αδειοδότησης θα περιληφθεί. Αυτή η ανάλυση θα ακολουθηθεί από νομοθετικές προτάσεις για την βελτίωση του βασικού κανονισμού βιολογικής καλλιέργειας. Το Ευρωκοινοβούλιο θα συμμετάσχει πλήρως στην βελτίωση αυτού του κανονισμού και στα κριτήρια βεβαίως αδειοδότησης των ουσιών που θα περιληφθούν στην βασική πράξη μετά από αυτή τη βελτίωση που προτείνουμε. Το Κοινοβούλιο λοιπόν θα συμμετάσχει διότι η μεταβολή του κανονισμού θα γίνει μέσω της κανονικής νομοθετικής οδού. Από τη στιγμή που θα έχουμε συζητήσει την ουσία και θα έχουμε συμφωνήσει και τα κριτήρια, νομίζω ότι τα διαδικαστικά θέματα που μας απασχολούν σήμερα θα είναι πολύ λιγότερο έντονα, διότι με την προσαρμογή του βασικού νομικού πλαισίου θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για τα πιο ε, για εξειδικευμένα κριτήρια αδειοδότησης. Και φαντάζομαι ότι τότε οι ανησυχίες σας θα αποδυναμωθούν. Συνοψίζοντας, μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαίρομαι για την πρότασή σας να υποβληθεί, να γίνει ψηφοφορία για την ευθυγράμμιση αύριο έτσι θα έχουμε την άποψη του Κοινοβουλίου και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις συζητήσεις τις διαθεσμικές πάνω σε σαφέστερη βάση. Και ελπίζω ότι γρήγορα θα οδηγηθούμε σε μια συμφωνία ε, χωρίς ε, ανησυχία. Επαναλαμβάνω ότι και εγώ ο ίδιος θα συμμετάσχω πλήρως σε αυτή τη φάση της τελικής συζήτησης και κάθε φορά που θα λαμβάνεται μία απόφαση που ενισχύει το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου σεβόμενοι ε, ταυτόχρονα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας και οι κανονισμοί που συζητούμε θα φροντίσω λέω ε, το Ευρωκοινοβούλιο πάντοτε να αναλαμβάνει ε, ενεργά το ρόλο του, του συνομοθέτη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ιωσήφ Μάτουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο συζητήτη της Περιφερειακής Επιτροπής συγχαίρω όλους τους συζητητέ για τα εξαιρετικά έγγραφα που κατέθεσαν στην κοινή αυτή συζήτηση. Οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολλές ε, προκλήσεις όπως ε, δημογραφική αποδυνάμωση, περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και ούτε καθεξής. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ένας απότερος στόχος, η βελτίωση δηλαδή της ανταγωνιστικότητας η βελτίωση των υποδομών και η ενίσχυση της διαφοροποίησης των περιφερειών. Υπό το φως αυτό και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως πρεσβεύω τα εξή. Πρέπει να βελτιωθεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την ε, τοπική ανάπτυξη. Με ένταξη των τοπικών εκπροσώπων στα εθνικά δίκτυα, με την δημιουργία online counseling, δηλαδή ε, χορήγηση συμβουλών στους γεωργούς μέσω διαδικτύου και τέλος συμβατότητα μεταξύ των ε, στόχων του ΦΕΝΤΕΡ και των στόχων της τοπικής συνοχής. Ονομάδων και ο εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνάδελφος κ. Χάνς Πέτα Μάγερ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνος είναι κρίσιμος συνομοθέτης. Έχει λοιπόν νέα δικαιώματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα οποία θα ασκήσει, οφείλει να ασκήσει. Εξ αυτού συμπεραίνω το εξής. Πρώτον, θα εργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα να τα ρυθμίσουμε με τις βασικές νομοθετικές πράξεις για να δώσουμε την μέγιστη δυνατή ασφάλεια σχεδιασμού στους αγρότες. Δεύτερο, θα καταβάλουμε προσπάθειες να δημιουργήσουμε και την απαραίτητη ευκαμψία μέσω των πράξεων εξουσιοδοτήσεως. Τρίτο, σε αιτιολογημένες μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις θα δώσουμε την δυνατότητα προσαρμογής τεχνικών λεπτομεριών μέσω εκτελεστικών πράξεων. Άρα, θα αγωνιστούμε υπέρ της διατήρησης και άσκησης των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων ως δημοκρατικά εκλογμένου οργάνου. Ζητώ από το Συμβούλιο να εγκαταλείψει την άκαμπτη στάση του και να, επι... να δεχθεί μάλλον τις κατεξουσιοδότησης πράξεις για ρυθμίσεις. Δεν πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις. Πρόκειται για τις αρμοδιότητες και την τήρησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της ε, S&D το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Ολέσνικα Τσακ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πολύ σημαντική συζήτηση, πολύ σημαντικές αποφάσεις. Είναι γεγονός ότι συζητούμε εδώ τεχνικές λύσεις, οι οποίες προκύπτουν ως αναγκαιότητα μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιε ρυθμίσει θα γίνουν με κατεξουσιοδότηση πράξη και ποιε με εκτελεστικέ. Στο μέλλον πώ θα ασκείται η κοινή αγροτική πολιτική. Θα συζητούμε περισσότερο για τι τεχνικέ πτυχέ ή για τα ουσιώδη περιεχόμενα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θέλει συγκεκριμένε λύσει. Αποδείξαμε στη συζήτηση ότι εμείς συμπαρατασσόμεθα με του αγρότε. Αγωνιζόμαστε υπέρ των άμεσων ενισχύσεων. Είμαστε οι σύμμαχοι των αγροτών ο μεγάλος ρόλος της συνθήκης της Λισαβόνας απηχείται στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δυνατόν να καταμετρηθούν ακριβώς πόσες θα είναι οι κατεξουσιοδότητες συμπράξεις και πόσες θα είναι οι αεκτελεστικές πράξεις. Δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση κύριε Επίτροπε, πρόκειται για την τήρηση και την εφαρμογή του δικαίου. Η απόφαση αυτή μπορεί πάντοτε βεβαίως να προσβληθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εάν ε, είναι μια τέτοια απόφαση αιτιολογημένη, δικαιολογημένη. Τότε βέβαια όμως θα αρθούν οι συνέπειες των πράξεων και δεν θα ωφεληθούν έτσι οι ε, αγρότες. Οι προτάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως ήταν καλά προετοιμασμένες. Συνάδελφος κύριο George Λάιον για δύο λεπτά. Uh, thank you, uh, President, uh, Commissioner. Uh, along with uh, my colleague... Ο Πάλο Δεκάστρο και άλλοι και εγώ ατυχώς συμμετέσχομεν σε διαπραγματεύσεις με Συμβούλιο και Κομισιόν για τον οριζόντιο κανονισμό επί 18 μήνες και με τρεις διαφορετικές προεδρίες και μέχρι σήμερα λίγη πρόοδος έχει επιτευχθεί παρόλες τις προσπάθειές μας. Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται η άποψη του Συμβουλίου ότι κάθε απόφαση για την ε, παράγωγη νομοθεσία θα πρέπει να γίνεται με εκτελεστικές πράξεις και όχι με εξουσιοδότηση. Βεβαίως από το Συμβούλιο δεν είναι κανείς εδώ να ακούσει. Οι εκτελεστικές πράξεις επιφυλάσσονται μοναχά για μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθεσίας. Ωστόσο, η θέση του Συμβουλίου φαίνεται πως είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να έχει λόγο καθόλου για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παραγωγή νομοθεσία. Δεν έχουμε λόγο. Αυτό λέει το Συμβουλίο. Δεν έχει αντιληφθεί όμως ότι η συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού και δεν μπορεί να συνεχιστεί business as usual. Η Κομισιόν σωστά λέει ότι είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Όμω, ξανά και ξανά στι διαπραγματεύσει για την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η ε, Κομισιόν συμπαρατάχθηκε με το Συμβούλιο και αρνείται έτσι τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Αντίθετα θα πρέπει να αγωνιστεί υπέρ των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου και υπέρ τη ορθή ερμηνεία των διατάξεων τη Λισαβόνα. Ακούω αυτά που λέτε σήμερα, ότι κατανοείτε δηλαδή το δίκαιο του αγώνα μας. Αλλά δεν συμβαδίζει με τις εμπειρίες που έχουμε, κύριε Επίτροπη, συλλέξει από τη μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων. Βγαίνει καθαρά από τη σημερινή συζήτηση ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να αγωνίζεται για να προστατεύσει τα δικαιώματά μας υπό τη συνθήκη της αγώνας, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πάρει όμοιρο την τελική απόφαση για τον κανονισμό μέχρι ότου συμφωνήσουν σε ένα λογικό συμβιβασμό Συμβούλιο και Επιτροπή για το ρόλο του Κοινοβουλίου ως συνομοθέτου. Ο συνάδελφος κύριος Νίκολσον έχει το ρόλο για δύο λεπτό. Thank you very much, President. Uh, while the issue of alignment of the Lisbon Treaty is maybe not the most riveting issue going through the committee at the moment, especially considering our work on the CAP reform. Όσον αφορά το έργο μας για την CAP Θέλω πραγματικά να συγχαρώ το έργο των εισηγητών. Ο φάκελος αυτός είναι πολύ περίπλοκος και με πολλές νομικές δυσκολίες το αναγνωρίζουμε αυτό. Δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε συμφωνία, όμως το θέμα πρέπει να προχωρήσει και αύριο θα έχουμε μια σαφή τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο κενό τώρα μεταξύ Κομισιόν και Ευρωκοινοβουλίου. Ε, υπάρχουν εξουσίες νέες στο Ευρωκοινοβούλιο βάσει της Λισαβόνας και τις υποστηρίζω. Όσον αφορά τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση, υποστηρίζω την ανάληψη εξουσίας και ελέγχου εκ μέρους του Κοινοβουλίου, γιατί είναι εκλεγμένα τα μέλη. Θέλω όμως το Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσει αυτές τις εξουσίες με την Προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας με σοφία και δημοκρατικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κολσον ε, και τελευταίο ομιλητής σε αυτή την κατηγορία εξ ονόματος της ομάδος EFD είναι ο συνάδελφος κύριος Άγνιου. Για 1,5 λεπτό. Well, the term implementing act is enough. Ο όρος εκτελεστική πράξη οδηγεί στα πιο βαθιά χασμουριτά. Αν όμως πει κανείς προσοχή, πάει η Κομισιόν να αρπάξει εδώ και άλλε αρμοδιότητε, τότε ο κροτισμός μου θα ξυπνήσει. Λίγο με εκπλήσει που η Κομισιόν σπρώχνει τα πράγματα στα άκρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε είναι, προσπαθεί απεγνωσμένα να αποφύγει τα δημοψηφίσματα. Εδώ ολοκληρώνουμε λοιπόν το εγχείρημα να γίνει αυτό. Και ένα από τα πράγματα αυτά είναι και για τη βιολογική γεωργία που είναι από τις πιο προστατευμένες βιομηχανίες σε ολόκληρη την ε, σε όλο τον κόσμο. Οι βιολογικοί γεωργοί έχουν αποκλειστικές, αποκλειστική πρόσβαση σε ορισμένες ενισχύσεις, εξαιρούνται από την ενόχληση των μέτρων πρασινίσματος που οφείλουν να υποστούν άλλοι ε, αγρότες και όμως παραμένουν πανάκριβοι. Σήμερα 3 Ιουλίου αυτός που φτιάχνει ζωοτροφές στη Μεγάλη Βρετανία έχει έξτρα δαπάνες για να έρθουν οι πρώτες ύλες στο εργοστάσιό του. Θα έπρεπε λοιπόν να φροντίσουν τις ανάγκες των πραγματικών γεωργών και όχι να παίζουν τους προστάτες των βιολογικών γεωργών οι ηθήνοντες. Πρώτος στο κατάλογο είναι ο συνάδελφος κ. Σιεκέρσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα περιστρέφεται γύρω από τι αρμοδιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ χρειάζονται ορισμένε προσαρμογέ. Στου κανονισμού, για παράδειγμα, πρέπει να διευκρινίζεται τι θα εκτελείται μέσω εκτελεστικών και τι θα γίνεται μέσω κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Άρθρα 290 και επόμενα. Αλλά δεν είναι τεχνικό το θέμα. Δεν είναι τεχνική η συζήτηση αυτή. Πρόκειται στην πραγματικότητα για αγώνα περί της εξουσίας ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα. Το άρθρο 43 παράγραφος 3 είναι ένα παράδειγμα του αγώνα αυτού. Νομίζω ότι τα πολύ σημαντικά πράγματα στην κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να ρυθμίζονται στον οριζόντιο κανονισμό. Μετά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Πρέπει όμως να εξετάσουμε προσεκτικά το ποιόν των κατεξουσιοδότησης πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων. Οι λεπτομέρειες εδώ έχουν μεγάλη σημασία. Γι' αυτό θα είναι καλό να υποβάλει πρόταση σχετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε θα πρέπει να είμαστε πλέον ενήμεροι, καλύτερα πληροφορημένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετέχουμε στις διαπραγματεύσεις και μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Στον τριμερή διάλογο κρίνονται τώρα όλα. Και όμως η τριμερή αυτή διάλογη δεν είναι ανοιχτή σε όλου, ενώ θα έπρεπε να είναι ανοιχτή σε όλου όσοι ενδιαφέρονται. Ο Επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφο κύριο Μάρκ Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, πριν να μιλήσουμε επί της ουσίας, να μιλήσουμε και για την τεχνική. Γιατί όπως είπε και πριν από μένα ο Παύλο Ντεκάστρο, Λάιον, Κάπουλα, Σάντος και άλλοι, το Συμβούλιο έχει τάση να αποφεύγει τις ε, ε κατεξοδότηση κάτι το οποίο περιορίζει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και είναι αντίθετο με τη συνθήκη αγώνας Μετά από τις πανεβάσεις που έγιναν στην Επιτροπή Γεωργίας, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώσει τις εξουσίες που μας ε, δίνει η συνθήκη. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι είναι η μοναδική ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτή της ΚΑΠ, διότι ε, εφαρμόζεται εδώ και 50 χρόνια και κινητοποιεί ένα τεράστιο ποσοστό του προπολογισμού. Θα πρέπει να υπάρξει επεξορρόπηση προ όφελο τη δημοκρατία, μεγαλύτερε αρμοδιότητε στο κοινοβούλιο. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε την παρακόλληση που δημιουργεί το Συμβούλιο αυτό η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και χαίρομαι για την θέση του Κοινοβουλίου και την απόφαση που θα πάρουμε αύριο. Άκουσα την άποψή σα, κύριε Επίτροπε, διότι σίγουρα σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είσαστε στο πλευρό μα προκειμένου να μπορέσει να εφαρμοστεί στην κλίση από Ευχαριστώ. Ο ομιλητή Ευχαριστώ, Πρόεδρε έκθεση του συναδέλφου με βρίσκει σύμφωνο σε ό,τι αφορά την ε, θέματα που αφορούν τη μείωση των ετησίων εκθέσεων ε, κλπ. Ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, οι διάφορες σύμβουλες και περιορισμό στο διοικητικό άκτου Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ντεκάστρο σχετικά με την ανάγκη να μην αποκλειστούν οι πληστή στήριξη στον τομέα των προκυπευτικών και τα μέτρα υπέρ της ε, ε, λειτουργίας των ενώσεων παραγωγών. Θεωρώ λοιπόν, όπως και ο εισηγητής, ότι τα κράτη-μέλη τα οποία συμφώνησαν με περιφερειακά προγράμματα ε, θα πρέπει να υπάρξει η αυτόματη αποδέσμευση των πόρων σε επίπεδο κράτους μέλους. Συμφωνώ και με την θέση του Κάπουλας Σάντος ε, για το ζήτημα της χρηματοδότησης ε, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγύηση. Συμφωνώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους για την εργασία τους. Δίνω τώρα το λόγο στη συνάδελφο κυρία Πατράο Νέβες Μαρία Ντοσέου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ως σκιώδης εισηγήτρια για την έκθεση σχετικά με την σήμαση και των βιολογικών προϊόντων. Να συγχαρώ τον συνάδελφο Χάουσλινγκ για τον τρόπο με τον οποίο μπόρεσε να διαχειριστεί το τριμμένο διάλογο αναφορικά με, τον με την ευθυγράμμιση γνώμη στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Σε ό,τι αφορά τα άρθρα 17 και 21, ζητήσαμε η αδειοδότηση ε, σε ό,τι φορά τις ουσίες να είναι μια ε, πράξη, ε, εκτελεστική πράξη και όχι κατεξοδότηση σύμφωνα με, τον, ε, με τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν αρχικά συμφωνούσε με το Κοινοβούλιο και το στήριζε, αλλά εν τέλει άλλαξε πορεία και στήριξε το Συμβούλιο. Τώρα υπάρχει και ο κατάλογος με τις ουσίες, αλλά τελικά απορρίφθηκε. έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουμε κατά νου την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει συνένεση, αλλά θα πρέπει να εκδηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας τόσο για το σήμερα όσο για το αύριο. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε την επίλυση του προβλήματος προσπεύοντας και στο ανώτατο... Κυρία Ελίζαμπεθ Κιώστιγκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, είναι μεγάλο κρίμα που παρόλου του τριμερείς διαλόγους λόγω των ανοιχτών οριζόντιων θεμάτων, δεν προέκυψε συμφωνία με το Συμβούλιο. Και μιλούμε για διαπραγματεύσεις οι οποίες έχουν διαρκέσει άνω του έτους και έχουν κοστίσει χρόνο και κόπο και που τελικώς απέστησαν του στόχου των. Ενώ αναφέρονται κυρίως στο τεχνικό μέρος μιας προσαρμογής ευθυγράμμισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας που είναι κέριος ωστόσο για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο, σημειώνω ένα πράγμα. Σε διαπραγματεύσει το Κοινοβούλιο έδειξε την συγκαταβατική του, συνενετική του διάθεση. Τέτοιο πράγμα δεν είδα από το Συμβούλιο όσο κατέστη καν δυνατόν να διαπραγματευτούμε, διότι από πλευρά Συμβουλίου δεν υπήρχε καν διαπραγματευτική εντολή. Δεν θέλω να προβώ σε υποθέσει, αλλά φαίνεται να πιστεύουν ότι η κέρυοι αυτή τομή για την τροποποίηση τη κοινή αγροτική πολιτική αναμένουν ότι το Κοινοβούλιο θα παραιτηθεί των θέσεών του, αλλά κάνουν λάθο, Θα προχωρήσουμε με ξεκάθαρη διαπραγματευτική εντολή στι διαπραγματεύσει για την τροποποίηση τη κοινή αγροτική πολιτική. Διοντές. Μεταβαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye και έχουμε μία δήλωση βουλήσεως. Δίνω το λόγο στην συνάδελφο κυρία Πρέντεργκάστ. Thank um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτές τις εκθέσεις απόψε, διότι ε, δείχνουν το σημαντικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Επιπτώσεις και ε, αποτελέσματα οι συζητήσεις αυτές έχουν για πολλούς πολίτες και έτσι οι εκπρόσωποι τους μπορούν να μιλήσουν εκ μέρους τους. Η συνθήκη της Λισαβόνας προέβλεπε μεγαλύτερο ρόλο για το θεσμό μας το Συμβούλιο και η Κομισιό μονίμως προσπαθούν να παρεκκλίνουν από αυτό και βεβαίω αυτό φαίνεται από τις πράξεις κατά εξουσιοδότης που γίνονται εκτελεστικές. Όπως και άλλοι ευρωβουλευτές είχα συναντήσεις δημόσιες με τους ενδιαφερόμενους στην περιφέρεια μου για την ΚΑΠ μετά το 2013. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες αλλά ελπίζουν ε, οι πολίτες της Ευρώπης ότι η νομοθεσία θα τους βοηθήσει. Γι' αυτό ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι σημαντικότατος. Κύριε Τσόλος, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις να υπογραμμίσω αυτό που ανέφερα στην ε, εισαγωγική μου ομιλία, ιδιαίτερα να απαντήσω τον κύριο Λάιεν ότι η Κομισιόν θα στηρίξει το Κοινοβούλιο κάθε φορά που αυτό θα καταστεί δυνατόν από νομική σκοπιά σύμφωνα με την διατύπωση και το περιεχόμενο των άρθρων 290 και 291. 290 που προβλέπει πως οι κατεξόδοτες πράξεις εφαρμόζονται στην περίπτωση όπου τροποποιούμε ή συμπληρώνουμε μη ουσιώδη ε, στοιχεία της, ε, ε, του βασικού άρθρου και το άρθρο 291 που όπως είπατε δίνει την δυνατότητα στην Κομισιόν να εξασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή των βασικών πράξεων το, μέσα σε αυτό το πνεύμα εργαστήκαμε και θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να βρούμε την τελική φόρμουλα και την επίτευξη συμφωνία. Ο κύριος Νίκολσον, ο οποίο όμως αναχώρησε, μίλησε για αυξανόμενες εντάσεις ανάμεσα στην Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Να σας διασφαλίσω ότι εγώ δεν πρόκειται να τροφοδοτήσω αυτές τις εντάσεις. Θεωρώ πως είναι προς το συμφέρον όλων και των γεωργών ιδιαίτερα, αλλά και των καταναλωτών Ευρωπαίων πολιτών να εξευρεθεί λύση. Τώρα, για τον κανονισμό για την οικολογική γεωργία, κυρία Πάτρας ε, ανεφέρθηκε. Είμαι έτοιμος ε, προς εξέβρεση λύσης ε, με εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία σχετικά με την απόφαση επί των ουσιών. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι και το συμφέρον των παραγωγών στην βιολογική γεωργία για να μην παρατείνουμε μια διαδικασία λήψη απο, από... απόφασης. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ στο πλαίσιο της προσαρμογής του βασικού κανονισμού για την ιδεολογική γεωργία να προβλέψουμε με τρόπο σαφή, περισσότερο από ό,τι τώρα τουλάχιστον, ποια είναι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εγκρίνουμε την ε, εισαγωγή μιας ουσίας και όταν τα κριτήρια αυτά θα καταστούν σαφέστερα και θα γίνει με βάση την ε, ε διαδικασία τότε η Κομισιόν θα ε, προτείνει εκτελεστικές πράξεις για να περιοριστεί ο ρόλος Κομισιόν στην εφαρμογή των κριτηρίων που θα συμπεριλαμβάνονται στα βασικά κριτήρια. Επίσης υπάρχει και η άλλη δυνατότητα που αναφέρεται να θέσουμε τον κατάλογο στο παράρτημα της ε, βασικής πράξης. Αλλά τότε για κάθε ουσία θα πρέπει να ακολουθούμε την ε, συνήθη τακτική τη συνήθεια διαδικασία, κάτι το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την υιοθέτηση. Αν συμφωνήσουμε λοιπόν με ένα πακέτο κριτηρίων ότι στην ε, βασική πράξη θα πρέπει να συμπεριφερθεί στις ουσίες, ίσως να κατορθώσουμε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να συμφωνήσει με την όλη αυτή τη διαδικασία. Προτείνω να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις επιλογές για να πετύχουμε ένα συμβιβασμό. Και στο πλαίσιο αυτού του συμβιβασμού θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Ευχαριστώ. Δευτερολογία εισηγητών, ο πρόεδρος κ. Παύλο Ντεκάστρο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Δράτω με αυτή τη ευκαιρία που μου δίνετε με το ένα λεπτό να ευχαρίσω τους συναδέλφους ε, και αλλά και τον Επίτροπο. Καταγράψαμε την, την στήριξη που μας έδωσε σήμερα ο Επίτροπος. Ε, ε, γιατί η ελπίδα εξέβρεση ε, συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τι εκτελεστικέ πράξει, δεν θα πρέπει να μεταφραστούν σε δυσκολία για την επίτευξη συμφωνία επί τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτικής. Γι' αυτό κάνω έκκληση προ τον Επίτροπε. Βρισκόμαστε στην εποχή τη Λισαβόνα. Χρειάζεται το Συμβούλιο να καταλάβει πω το Κοινοβούλιο έχει νέε αρμοδιότητε, νέε εξουσίε και δεν προτίθεται να παρετηθεί από αυτές. Αύριο με την ψήφο Επίτροπε, εμεί θα ακολουθήσουμε την θέση τη Κομισιόν και ελπίζουμε πω ε, τόσο και το Συμβούλιο στο τέλο να ευθυγραμμιστεί με τι θέσει αυτέ. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ηγητή, ο κύριος Τζοβάνι Λαβία, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως η συζήτηση ήταν χρήσιμη, εν πάση περιπτώσει διότι μετά από τα όσα αδελφοί σχετικά με τις θέσεις τους για την επιγράμμιση της αγώνες μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία του Επιτρόπου πως το Κοινοβούλιο επιθυμεί να διατηρήσει τον ρόλο του και τις αρμοδιότητές του. Είναι σαφές λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πέραν των αποτελεσμάτων της αυνής ψηφοφορίας που δεν νομίζω ότι ουσιαστικά θα διαφέρει από τις θέσεις που αρχικά είχε διατυπώσει η Κομισιόν, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και το δρόμο πρέπει να διανύσουμε, όχι μόνο σε ό,τι φορά την εφαρμογή των ε, αρμοδιοτήτων που μας παρέχει η Λισαβόν αλλά και την εφαρμογή της ε, νέας αγροτικής πολιτικής επίτροπε. Ξέρετε πολύ καλά πόσες φορές συναντηθήκαμε ε, κάτω από διάφορες προεδρίες γνωρίζετε πολύ καλά που πως κολλήσαμε σε κάποια ζητήματα οριζόντιας φύσης και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε και μας κόστισε τόσο σε ό,τι φορά τον χρόνο που χρειάστηκε, τι προσπάθειε που καταβάλαμε κλπ. Πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι αυτόν τον δρόμο. Αύριο είναι μια ενδιάμεση φάση όπου το Κοινοβούλιο θέλει για μια ακόμα φορά να εκφράσει με σαφήνεια την θέση του και την βούληση να μην παρτιθεί από τι αρμοδιότητες ή τις εξουσίες. Αλλά χρειάζεται να ξεκινήσουμε τη δουλειά διότι ε, ευθυγράμμιση προς τη συνδίκη της Λισαβόνας ε, και η καθυστέρηση αυτή δεν θα πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδι. σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική μεταρρύθμιση αυτή, ε, θα, ξα... θα ξαναπούμε, θα συναντηθούμε κλπ. Αλλά για το ζήτημα τη ευθυγράμμιση τη δική τη Λισαβόνα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να επιταχύνουμε. Συνάδελφο κύριο Μάρτιν Χόισλινγκ, που έχει το λόγο για δύο λεπτά. <clears throat> Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ και πάλι για την συμβιβαστική διάθεση που δείξατε. Καθιστώ σαφές ότι από πλευρά Κοινοβουλίου δεν είναι μια στήρα αιμονή σε κάποιες αρχές, αλλά πρόκειται για μια προσπάθεια ρύθμισης για το μέλλον που θα πρέπει να ισχύει για όλους, και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δεν μπορούμε να δεχθούμε συμβασμούς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να σταθούν στο μέλλον. Πρέπει να, στερεο, να στεκόμαστε σε στέρεο έδαφος για χρόνια. Καμιά φορά βρίσκω ότι είναι έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Καμιά φορά και από πλευρά Συμβουλίου απέναντι στο Κοινοβούλιο. Το είπατε κι εσείς εμέσως ότι ενδεχομένως καθυστερούν με τον τρόπο αυτό τα διαφορά νομοθετήματα. Ναι, ίσως υπάρξουν, σημειωθούν κάποιες καθυστερήσεις από την άλλη μεριά δεν μπορείτε να στερηθείτε την ε, εμπειρογνωμοσύνη του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, προτείναμε να περιληφθούν οι ουσίε στον βασικό κανονισμό, γνωρίζοντας ότι, θα, ότι υπήρξαν μάλλον δύο αλλαγέ μέσα σε μια τετραετία που μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν με ταχύε διαδικασίε και από πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν αντιμετωπιστεί με ταχύε διαδικασίες ενώ μάλλον το Συμβούλιο φοβάται ότι το Κοινοβούλιο θα προκαλεί καθυστέρηση. Όμως αυτή η φόβη είναι σαφώς αδικαιολόγητη. Εμείς θα επιμείνουμε στα δικαιώματά μας. Και νομίζω το μήνυμα αυτό πρέπει να το λάβει και το Συμβούλιο, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε οτιδήποτε, ούτε να δεχθούμε συμβασμούς οι οποίοι δεν μπορούν να σταθούν. Πρέπει να είναι ένας έντιμος πολιτικός διάλογος μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ που θέσατε και πάλι, α, εκδηλώσατε μάλλον τη διάθεση να υποβάλλετε συμβαστικές προτάσεις. Πιστεύω ότι με τέτοια βήματα θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τον κανονισμό με τρόπον ώστε να συμφωνήσουν όλοι. Αυτό που θέλουμε εμείς ως Κοινοβούλιο είναι να προχωρήσουμε ταχαίως σε διαδικασίες που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι το Κοινοβούλιο μπλοκάρει την περαιτέρω πρόοδο. Αυτό δεν το θέλουμε με κανένα τρόπο. Θέλουμε όμως ένα πλαίσιο το οποίο να εξυπηρετεί, να σέβεται και τα δικά μας συμφέροντα και δικαιώματα. Θα το πω καθαρά. Συμβιβαστική διάθεση έχει δείξει μέχρι τώρα μόνο το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο όχι, σπάνια. Με την δευτερολογία του εισηγητού κυρίου Καπούλα Σάντος. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως όλα υπόθηκαν. Έχω ελάχιστα να προσθέσω. Να πω ότι τα σημεία που μόλις συζητήσαμε καταδεικνύουν με τρόπο σαφή ότι υπάρχει συνεκτική θέση του Κοινοβουλίου και επιθυμούμε την εξέβριση μιας συμφωνίας. Είμαι βέβαιος πως η Κομισιόν θα δεσμευτεί προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω το αυτό να συμβεί το συντομότερο. Συνάδελφοι, η κοινή συζήτηση που είχε στο επίκεντρο κρίσιμες πτυχές της διαθεσμικής συνεργασίας έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30 πέρας εργασιών για σήμερα.